να να εθετήσουν δεσμευτικούς στόχους γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον Επίτροπο. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η προφορική ερώτηση στην Επιτροπή είναι και της εποχής για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Εισηγείται και πάλι η κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, οδηγία για τα παιχνίδια. Είχαμε τον εξή στόχο, να καθεστήσουμε πιο ασφαλή τα παιδικά παιχνίδια, γιατί παιχνίδια τα οποία βρίσκονται ακριβώ πάνω στην εξέλιξή τους, αντιδρούν ιδιαίτερως ευαίσθητα σε επικίνδυνε χημικές και τοξικές ουσίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα τότε ε, έγκυρα επιστημονικά στοιχεία ε, διατυπώσαμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ε, ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως το θέμα αυτό το εξετάζουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και για μένα ως μητέρα το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό να έχουμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί υπάρχουν νέες ε, ε, μελέτες που δείχνουν ότι τα ανώτατα κατόφλια για τα βαρέα μέταλλα δεν είναι αρκετά αυστηρά και συμπεριλάβαμε μία ρήτρα στην οδηγία η οποία επιτρέπει την εκ των υστέρων ε, διόρθωση των ανώτατων ορίων. Και νομίζω θα πρέπει να κάνουμε χρήση αυτή της ρήτρα. Ε, κύριε Ταγιάννη, ε, είχαμε ευθυνθεί τον προκάτοχό ήδη πριν από ένα χρόνο. Ε, χαίρομαι που η Επιτροπή πρόκειται να εξαγγείλει ότι τα νότατα όρια, τουλάχιστον για ορισμένα βαρέα μέταλλα, θα γίνουν αυστηρότερα. Νομίζω θα πρέπει εν γέν να εξετάσουμε όλες τι επικίνδυνε τοξικές ουσίες και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα βαρέα μέταλλα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις τοξικές ε, ουσίες, με τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάφρακες για παράδειγμα, τους ώστε ε, να υπάρξει εδώ μια βελτίωση, γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάθε χρόνο πάλι και πάλι κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την ασφάλεια των παιχνιδιών και κάθε χρόνο διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εδώ πολλές ελλείψεις. Και εδώ το διακύβημα είναι αυτές οι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες που είναι ιδιαίτερως επικίνδυνες για την υγεία των παιδιών και οι νέες επιστημονικές ε, γνώσεις Μα λένε ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να προσαρμοστούν σχετικά οι ωριακέ τιμέ. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλου να ασχοληθεί με αυτέ τι ωριακέ τιμέ. Και ε, χαίρομαι πάρα πολύ που προτίθεσε να το πράξετε κύριε Επίτροπε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το προβλήμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η παρακολούθηση τη αγορά. Και εδώ καλούνται οι χώρε μέλη να λάβουν τι ευθύνε του και να μεριμνήσουν ούτω ώστε να ε, βγαίνουν στην αγορά μόνο τέτοια παιχνίδια τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφαλείες. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε και αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τρίτο και τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να φέρω εδώ, ε, εδώ ε, ε, το ζητούμενο επίσης και σήμανση των παιχνιδιών. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι παρα... θεωρούν εσφαλμένα ότι η σήμανση η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι μια σήμανση ασφαλείας, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Σήμανση Ασφαλείας που να είναι πραγματικά αξιόπιστη και να μπορεί να ελέγχεται από ανεξάρτητες αρχές ή υπηρεσίες ούτω ώστε να μην μπορεί να συμβεί επικίνδυνα παιχνίδια να φτάνουν, να καταλήγουν στα ράφια των εμπορικών καταστημάτων ε, απειλώντας την υγεία των παιδιών μας. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κατεπηγόντως κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ασφάλεια των παιχνιδιών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όχι επειδή έχουμε φτάσει στην εποχή του χρόνου που αυξάνονται οι πωλήσει παιχνιδιών σε μεγάλο βαθμό. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι ότι υπάρχει απόλυτη προστασία των παιδιών και των καταναλωτών. Η αναθεωρημένη οδηγία έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα παιχνίδια που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρήση χημικών ουσιών. Τα μέτρα επιτήρησης αγοράς έχουν ενισχυθεί τα ε, στοιχεία, τα έγγραφα που πρέπει να έχουν διαθέσιμα οι κατασκευαστές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες της κατασκευής ε, των παιχνιδιών, τις ουσίες, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζουν αυτά τα παιχνίδια διαβάζοντας ε, την ε, επιστημονική γνωμοδότηση επιστημονικής ε, επιτροπής για την αξιολόγηση των ορίων μετανάστευσης διαπίστωσα ότι η μέθοδος μέτρησης της μετανάστευσης για χημικά στοιχεία στα παιχνίδια δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη. Χρειάζεται λοιπόν προσδιορισμός μιας μεθόδου μέτρησης για τις οργανικές καρκινογόνες, μεταλλοξιογόνες και τοξικές ουσίες και κυρίως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να δοκιμάζονται με ανεξάρτητο τρόπο. Οι τελευταίε εκθέσει RAPEX αναφέρουν ε, ε, κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την εποπτεία τη αγορά παιχνιδιών. Φτάνουν νέα παιχνίδια στην αγορά που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την πιο ευάλωτη ομάδα καταναλωτών. Η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να ενισχυθεί, είναι σαφέ αυτό, να εξασφαλιστεί το υψηλό, το, ο ψηλότερο βαθμό προστασία για όλα τα παιδιά. Πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην υπάρξουν κενά ή παραθυράκια για την κατά την εφαρμογή τη αναθεωρημένη οδηγία. Πρέπει κύριο στόχο μα να είναι η υποπτία τη αγορά, η, και, η, ανάλυση, και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περιέχουν τα παιχνίδια αυτά ε, επικίνδυνες ουσίες για τα παιδιά. Ο κ. Χάρμπορ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σπουδαιότητα της ερώτησης που υποβάλλουμε σήμερα οφείλεται στο ότι η Επιτροπή μας συνεχίζει να επαγρυπνεί ιδιαίτερα για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως και για όλα τα κατανοητικά αγαθά άλλωστε. Δώσαμε, λοιπόν μεγάλη προσπάθεια για να υιοθετήσουμε το 2009 την αναφερμένη οδηγία τα παιχνίδια. Τα πράγματα όμως δεν σταματούν εκεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ευπρόσδεκτο το ότι δίνουμε στην Επιτροπή και σε εμά την ευκαιρία να επανα να επαναδιαβεβαιώσετε ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, τις δοκιμές και να εξασφαλίσετε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία και η επερχόμενη νομοθεσία θα συνεχίσει να αναθεωρείται μόνιμα, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει την αύξηση των επιστημονικών στοιχείων για τα πιθανά επικίνδυνα χημικά στοιχεία. Αυτό περιλαμβάνει βέβαια και την ανάγκη μονίμων ε, μεθόδων ε, δοκιμών. Πολλές φορές ε, διαπιστώνουμε ότι οι κατασκευαστές παιχνιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να υπάρχουν στάνταρ πρότυπα, μόνιμα πρότυπα που πρέπει να τηρούν. Υπάρχει όμως και ένα εκτενέστερο θέμα. Το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η νομοθετική αντιμετώπιση, αλλά ολόκληρη η αλυσίδα προσφοράς των παιχνιδιών. Πολλά από αυτά έρχονται εκτός, από χώρε εκτός της Ένωσης. Πρόσφατα, ο συνάδελφός σας, κύριος Ντάλ, με κάλεσε να εκπροσωπήσω την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς σε μία μείζωνα τριμερή σύνοδο κορυφής ε, είπα Ένωσης και Κίνες να μιλήσουμε για θέματα ασφάλειας παιχνιδιών. Και ένα από τα σημαντικά ζητήματα που έκανε η Επιτροπή, ο κ. Ντάλη, και πραγματικά τον συγχαίρω γι' αυτό, είναι να δείξει σε κατασκευαστές με δύο της Κίνας ε, στοιχεία και ε, να τους μάθει το σχεδιασμό εξ αρχής των παιχνιδιών με βάση την, ε, τη, την τήρηση των δοκιμών. Άρα πρέπει να μεταφέρουμε τεχνογνωσία για να έχουμε ασφαλή προϊόντα από το ξεκίνημά τους. Τα προϊόντα αυτά κατόπιν πρέπει να τηρούνται, να, να συνεχίζονται με σωστά συστήματα δοκιμών. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Το θέμα δεν είναι μόνο η σήμανση, αλλά ούτε καν το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά όλοι στην αλυσίδα της ε, ε παροχής των προϊόντων να καταλάβουν τις ευθύνες τους. Η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σε αυτά που είπε ο κύριος Χάρμπορ. Όλα αυτά έχουν πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι εμεί θα πρέπει να κάνουμε, να λάβουμε ήδη τα καθήκοντά μας. Δεν είναι σύμπτωση κάθε φορά πριν από τα Χριστούγεννα και φέτος το ίδιο ε, θέτουμε το ζήτημα της ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών. Και πέρσι ήταν κυρίω οι καρκινογόνες ε, ουσίες ε, στα παιδικά παιχνίδια μας απασχόλησαν. Και ο Επίτροπος κ. Βερχόγγεν μας είπε ότι θα υπάρξουν νέες επιστημονικές ε, μελέτες. Οι επιστημονικές έρευνες έγιναν και οι οριακές ε, τιμές για τους ε, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες είναι εξαιρετικά υψηλές. Ε, αλλά και οι δοκιμές που γίνονται δεν είναι αξιόπιστες. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο ε, πώς θα προκυνήσει το θέμα και σε τι είδους κριτική θα καταλήξει εκείνο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιεκτικότητα σε μόλιβδο ε, οι τιμές ε, δεν είναι πλέον οι ενδεδειγμένες. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας θα προβλέψουμε άλλες οριακές τιμές για το μόλιβδο ή άλλα βαριά μέταλλα. Ε, επίσης αναμένουμε τις οριακές τιμές ε, για κατόφλια θορύβου που επιβαρύνουν την υγεία των παιδιών. Αυτό συζητήθηκε ήδη σε πρώτη ανάγνωση ε, και ελπίζω θα δεθεί ε, σύντομα το θέμα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το ζήτημα της εποπτείας της αγοράς, γιατί ακόμα και οι καλύτερες οδηγίες ε, δεν μπορούν να διατηρήσουν την αξία τους παρά μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής εποπτεία της αγοράς. Τέλος, το θέμα του τελωνίου. Και ξέρει ο κύριο ε, Ταγιάννη ότι, ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί, τους, μαζί του. Η κυρία Σάλντε Μόζε ως εισηγήτρια ε, θέλει να φροντίσει να γίνουν παραπέρα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα ε, παράλληλα με τις ορικέ τιμέ για τα βαριά μέταλλα και τι καρκινογόνες ουσίες. Ο κύριος Ταγιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση στην Ολομέλεια για την ασφάλεια των παιχνιδιών στην Ένωση δεν είχε ποτέ γίνει πιο, σε πιο επίκαιρη στιγμή, ιδίω με δεδομένο ότι πριν από λίγο καιρό το χώρε όπω το Βέλγιο πέσει από την αγορά μια σειρά προϊόντων, μια σειρά παιχνιδιών λόγω ε, συγκέντρωσης φορμαμίδης ενός καρκινογόνου μεταξιογόνου και τοξικού προϊόντος σε, σε επίπεδο που θεωρείται πλέον επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Και άλλες χώρες όπως η Γαλλία για παράδειγμα αύξησαν το επίπεδο επακρύπνησης για την εποπτεία της αγοράς σε ό,τι αφορά τα ίδια προϊόντα. Εμείς περιμένουμε την επίσημη κοινοποίηση των μέτρων που υιοθετούν οι εθνικές αρχές και κατόπιν θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των στοιχείων βάσει των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών μας. Αν βάσει των ελέγχων αυτών επιβεβαιωθεί βάσει επιστημονικών δεδομένων ότι όντω μια τέτοια συγκέντρωση φορμαμίδης αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των παιδιών, θα αναλάβουμε θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να τροποποιήσουμε μέσω διαδικασία επιτροπολογία τι διατάξει τη οδηγία προ την κατεύθυνση αυτή. Η οδηγία θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Χάρμπορ, προβλέπει αυτό το μηχανισμό που επιτρέπει να ενημερώνεται καθημερινά βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, ήδη ε, προέβη σε μια σειρά αλλαγών για διάφορες χημικές ουσίες που όπως ε, ανέφερε η κυρία Βάις Γκέρμπερ μεταξύ των οποίων ε, μόλιβδος και δμιο για να προσεγγίσει την, τα νότια στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Οι αλλαγέ αυτέ ε, θα υλοποιηθούν βάσει τη υφιστάμενη ε, ε, διαδικασία κανονιστική επιτροπή. Δεσμεύομαι τώρα να της κυρίας Ρουλή προσωπικά να διαφυλάξω, να διατηρήσω πλήρως την ενημέρωση του Κοινοβουλίου για τις εργασίες ε, και την εξέλιξή τους ό,τι αφορά τις δύο αυτές ουσίες. Για τα άλλα συγκεκριμένα ερωτήματα που είναι στο κέντρο των, ε, της προφορικής ερώτησης που υποβάλλατε, ξεκινώ με την ε, Επιστημονική Επιτροπή Κινδύνων για την Υγεία και το Περιβάλλον που παραπέμπει σε μια μελέτη του, του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την αξιολόγηση της μεθόδου που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια για τον εντοπισμό ίχνων βαρέων ε, μετάλλων ε, στα παιχνίδια. Η ανάλυση, η ανάλυση αυτή έγινε βάσει του κανόνα 1.71.3. Σύμφωνα με τη μελέτη, 40 εργαστήρια μετέσχαν στον έργο αυτό, 15 από αυτοί είναι οργανισμοί πιστοποιημένοι από τα κράτη-μέλη ως ε, ικανά να εξετάζουν την, συμφων... την συμμόρφωση των παιχνιδιών στην οδηγία. Μόνο τρία από τα 40 εργαστήρια ερμήνευσαν με, εσφαλμένο τρόπο τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη, διορθονομιλητής, που ενώ δόθηκαν για τα ονόματα των εργαστηρίων και κλήθηκαν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τα σκόπιμα μέτρα. Επίση, τα αποτελέσματα τη μελέτη δόθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστοποίηση για να λάβει υπόψη στα πλαίσια τη αναθεώρηση των σχετικών κανόν, του κανόνα EN713 που ισχύει αυτή τη στιγμή, με στόχο την υιοθέτηση νέου προτύπου μέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται για την εφαρμογή των νέων διατάξεων σχετικά με τι χημικέ ουσίε, δηλαδή το 2013. Σε ό,τι αφορά τη νέα οδηγία για τα παιχνίδια που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2009, η οδηγία αυτή τηρεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση του εμπόριου των προϊόντων και προβλέπει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και εποπτεία τη αγορά. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία για να εξασφαλίζουν ότι μόνο τα ασφαλή προϊόντα θα φτάνουν στα χέρια του Ευρωπαϊκού Καταναλωστή. Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο την ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα, όσο και την αποτελεσματική, αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης των προϊόντων που βρίσκονται ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε μια περίπτωση εν τέλει που τα κάτι μέλη αντιμετωπίσουν παρατυπίες στα παιχνίδια είναι σημαντικό να κοινοποιούν αμέσως την πληροφορία αυτή σε στα άλλα κράτη-μέλη μέσω του ΡΑΠΕΞ, του Κοινοτικού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών ε, με ταχύ τρόπο. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις κινέζικες ιδίως αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών, κύριε Χάρμπορ. Η Ευρωπαϊκή οι εμπειρογνώμονε από την Ευρώπη και την Κίνα συναντιούν τακτικά και ανταλλάσσουν πληροφορίε για την νομοθεσία και τα πρότυπα που εφαρμόζονται, αλλά και για την διοικητική πρακτική σχετικά. Το προσωπικό των κινέζικων ερχών ε, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για να βελτιώσουν τον έλεγχο και την ποιότητα του ελέγχου στα προϊόντα αυτά. Σε ό,τι αφορά τα όρια χημικών ουσιών κύριε Μπουζόη προφανώς είναι να καλύτερο να υιοθετήσουμε μια μέθοδο που βασίζεται στη μετανάστευση γιατί εκτίθεται στην πραγματική, τον, εξετάζει τον πραγματικό κίνδυνο του παιδιού αλλά η αξιολόγηση των ορίων μετανάστευσης περιλαμβάνει και την κίνδυνο και την έκθεση σε, και σε κίνδυνο ε, για τον υπολογισμό και δυσκολεύει τον υπολογισμό των ε, ποσοστών. Επειδή οι χημικές ουσίες είναι κάμποσες πάνω από χίλιες και δεν έχουμε επαρκείς ε, πληροφορίες για όλες αυτές τις ουσίες, η μέθοδος αυτή, τη, στη φάση αυτή των επιστημονικών γνώσεων είναι αδύνατη. Βεβαίω η οδηγία προβλέπει ήδη όρια που βασίζονται στην μετανάστευση για κάποιες χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και επιτρέπει πάντα χάρη στην επιτροπολογία να μπορούμε να εισάγουμε στο μέλλον όρια που βασίζονται στη μετανάστευση σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμα περαιτέρω μεταγενέστερα στοιχεία για νέες ουσίες. Σε ό,τι αφορά τα, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονοάνθρακες, κυρία Ρούλε, ουσίες αυτέ βρίσκονται σε πολλά καταναλωτικά εργαλεία, ε, προϊόντα, όχι μόνο σε παιχνίδια. Δεν είναι λοιπόν... Ε, μάλλον ο έλεγχος αυτός ε, δεν γίνεται λοιπόν στα, μέσω της οδηγίας των παιχνιδιών αλλά μέσω του REACH που έχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής και αυτή η μέθοδος είναι και πιο αποτελεσματική και πιο συνεπής. Τα παιχνίδια για παιδιά κάτω των τριών ετών υπόκεινται σε πιο αυστηρούς κανόνες. Τα παιδιά, τα νήπια, είναι πιο ευάλωτα και χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ηλικία ε, χρήσης ενός παιχνιδιού, ο, ο παρασκευαστής πρέπει να υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνε, Ωστόσο, δεν θεωρούμε δικαιολογημένο να βάλουμε όλα τα παιχνίδια στου, ίδιους, περιορισμού με τα πολύ μικρά παιδιά. Η έκθεση των κίνδυνων και η χρήση τους δεν είναι πάντα ίδια. Επιπλέον, μια πλήρη απαγορεύση κάποιων προϊόντων για μεγαλύτερα παιδιά, για τα οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι προβλήματα θα ήταν κάτι δυσανάλογο και αντίθετο με τον στόχο της καλύτερης νομοθεσίας. Η νέα οδηγία ε, μιλά και για τις ε, κατηγορίες που υπάγονται, που χαρακτηρίζονται CMR, αλλά εδώ αποφασίστηκε ότι η πλήρης απαγόρευση χωρίς δυνατότητα παρέκκλησης δεν θα ήταν ούτε δικαιολογημένο ούτε και ρεαλιστικό αν η ουσία δεν παρουσιάζει προβλήματα στην υγεία, διότι είναι απροσπέλαστη για παράδειγμα, δεν μπορεί να απαγορευτεί. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται αναπερίπτωση ε, βάσει επιστημονικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα για κάθε ουσία. Μπορούν να υιοθετηθούν αυστηρότερα όρια μέσω της επιτροπολογίας για να εξασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. Η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική πρόταση οποτεδήποτε ο πραγματικό κίνδυνος και συγκεκριμένα δεδομένα το καθιστούν σκόπιμο. Όπως ξέρετε η νέα οδηγία θα είναι εφαρμοστέα για τους, ε, οικονομικούς, για επιχειρηματίες από του χρόνου τον Ιούνιο. Οι σχετικές υποχρεώσεις θα είναι εφαρμοστές λοιπόν από τον Ιούλιο του 2013. Για την Επιτροπή η εφαρμογή των νέων κανόνων από πλευρά όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κράτων, μελών και, και επιχειρήσεων αλλά και η ενσωμάτωση των προσαρμογών ε, της επιστημονικής νέας γνώσης αποτελούν προτεραιότητα. Ιδίω τα κράτη-μέλη ήδη συναντήθηκαν δύο φορές για να συζητήσουν τις τροποποίησει σε κάποιες υποχρεώσεις που αφορούν χημικές ουσίες τον Οκτώβριο του 2009 και τον Σεπτέμβριο φέτος. Προβλέπεται μια νέα συνάντηση τον Απρίλιο του χρόνου για να κλείσουν οι εργασίες. Η Επιτροπή στην Επιτροπή δημιουργήθηκε και μια μεικτή επιτροπή ειδικών για χημικά θέματα που συναντήθηκε τον Νοέμβριο με καλά αποτελέσματα για τον, και ασχολήθηκε με τον θορισμό, ορισμό των ζητημάτων που πρέπει να, επιλέγ, ασχοληθεί και των επιλογών που υπάρχουν. Μια νέα συνάντηση προβλέπει τον, τον Ιανουάριο του 2011. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς κύριε Χάρμπουρ, ε, στην δεύτερη απάντησή μου θα σας δώσω σχετικά, ε, τις απαντήσεις σχετικά στις ερωτήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόμη, πρόεδρε, η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος για την προστασία των παιδιών ε, μέχρι τα 14 καθορίζει τους βασι, τις βασικές απαιτήσει που πρέπει να τηρούν τα παιχνίδια όταν κατασκευάζονται και πριν μπουν στην αγορά. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίηση ε, επεξεργάστηκαν μια σειρά ευρωπαϊκών εναρμονισμένων κανόνων βάσει ε, κυρίων βασικών απαιτήσεων. Η αξιολόγηση τη συμμόρφωση των ε, παιχνιδιών εξασφαλίζεται από το σήμα CE που είναι υψηλό επίπεδο ασφάλεια σε σχέση με τα διεθνή στάνταρτ. Προφανώς έχω βεβαιότητα ότι έγκαιρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μικροτσίπ αντί για το σήμα CE. Θεωρώ προσωπικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεσμεύεται σε μόνιμη βάση για να ενημερώνει τις δοκιμές ασφάλειας, καθιστώντας πάντα συμβατές με τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο πρέπει να εκφράσω την ανησυχία μου, διότι ακριβώς στην περίοδο Χριστουγέννων συζητούμε μία μελέτη όπου γίνεται λόγος για μη συμμόρφωση των δοκιμών ε, για τα όρια της μετανάστευσης χημικών ε, στοιχείων των παιχνιδιών δεν χρειάζεται να, δεν πρέπει να δημιουργούμε ε, ανησυχίες βασιζόμενοι ε, στην ε, συνεχή ενημέρωση των δοκιμών, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δουλεύουν στον τομέα, στον κλάδο, τηρώντας όλες τις, όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι η βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από βελτίωση της εφαρμογής της. Ενώ η εργασία μας εδώ στο Κοινοβούλιο συνεχίζεται πάντα προς την κατεύθυνση της αύξησης της ποιότητας των παιχνιδιών. Η ευχή μου για το νέο έτος είναι οι μη ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν και αυτές, να, να υιοθετήσουν και αυτές το παράδειγμα των δικών μας στάνταρ, βελτιώντας την ποιότητα των δικών τους ε, προϊόντων. Ευχαριστώ. Η κυρία Πέρες. Δύο λεπτά. Presidente, comisario, ε, πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η, Επιτροπή, η οδηγία που εγκρίθηκε το 2009 είναι μια επιτυχία γιατί ανανεώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφαλεία των παιχνιδιών. Είναι ένα μεγάλο βήμα στη σωστή κατεύθυνση γιατί σηματοδοτεί το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να, είμαστε, να επαγρυπνούμε πάντοτε σε σχέση με τα παιχνίδια τα οποία βγαίνουν στο εμπόριο τους ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιχνιδιών. Όλα τα παιχνίδια που βρίσκονται στην αγορά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς επαγρύπνησης για να ανοιχνεύσουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια ε, για τις λεγόμενες ε, τοξικές ουσίες, καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες κλπ και ε, άλλε επικίνδυνε ουσίε όπω είναι η πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακε. Είναι αναγκαίο ε, οι κανόνε που θα ακολουθούμε να είναι πιο ξεκάθαροι όσον αφορά τα ανώτατα όρια και τους ε, κινδύνους που προέρχονται από μια κατάλληλη χρήση. Θα πρέπει να πετύχουμε η ηλικία που συνιστάται για τα παιχνίδια να βασίζεται σε μελέτες συμπεριφοράς των παιδιών. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τους ε, κανόνες, τις ε, επιστημονικές προόδους που εδραώνονται σε σωστές έρευνες και να είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά την επαγρύπνηση στην αγορά και την ε, εισαγωγή των παιχνιδιών. Είναι αναγκαίο να συνεργαζόμαστε και να ενισχύουμε την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και να ε, συνεργαζόμαστε και με τα τελωνία όσον αφορά την εισαγωγή παιχνιδιών. Οι πολίτες θέλουν να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους και θα πρέπει να τους δώσουμε την ασφάλεια ότι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτοβα. Κύριε Επίτροπε, τα συμπεράσματα της Επιστημονικής Επιτροπής για τα όρια των έξι χημικών ουσιών δεν είναι απόλυτα αξιόπιστε. Γι' αυτό σας υποβάλλω το εξής ερώτημα. Συμφωνώ με τους εμπειρογνώμονες που είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί η ζημιά που προκαλούν αυτές οι ουσίες στα παιδιά, διότι στην προσημείωση χρησιμοποίησαν νερό και όχι το σύελο των παιδιών που έχει λακτόζη. Αλλά δεν πρέπει να επικρατήσει βεβαιότητα όταν μιλάμε για μικρά παιδιά και τους κινδύνους ε, που ε, ε, συνεπάγονται για αυτά τα πλαστικά παιχνίδια. Πρόκειται λοιπόν να κάνετε μια δοκιμή πάνω σε ποντίκια για να αναλύσετε τα, τις, τις, τις συνέπειες της χρήσης μπιφενόλης στα μπιμπερό που έχουν απαγορευτεί από το Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία προβλέπει έκθεση των παιδιών μέχρι 50% της έκθεσης που ισχύει για τους ενήλικες. Επειδή η Επιστημονική Επιτροπή θέλει να μειώσει τα όρια καδμίου σε 0,36 μικρογραμμάρια, θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής όσον αφορά τα μέτρα που θα ισχύσουν για τα παιχνίδια. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να μας δώσετε προθεσμίες για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς ποια θα είναι η κατάσταση ώστε να ενημερώσουμε τα παιδιά και τους γονείς τους. Κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε ε, λοιπόν καθώς άκουσα τον κύριο επίτροπο να μιλάει με τόση άνεση για τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες για τις καρκινογόνες και τοξικές ουσίες για μια στιγμή νόμισα ότι ήταν χημικός και όχι επίτροπος. μετά θυμήθηκα ότι είναι επίτροπος αρμόδιος για το θέμα άρα το πρώτο για το οποίο έπρεπε να μας απαντήσει με λεπτομέρειες ήταν για το σήμα ce το θέμα που έθεσε η εξαίρετη συνάδελφος evelyn Γκέπχαρτ, το σήμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι η εγγύηση ασφάλειας για τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά μας. μετά όμως σκέφτηκα πάλι ότι δεν απάντησε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο είναι δύο χρόνια ακριβώς σήμερα ή μάλλον την παρασκευή από όταν η πρώην επίτροπος της προηγούμενης κομισιόν υπέγραφε σε ένα μαγαζί παιχνιδιών σε ένα κατάστημα παιχνιδιών έξω από τις βρυξέλλες ένα σύμφωνο ασφάλειας με τους εμπόρους λιανικής αγοράς με τους λιανεμπόρους και τους εισαγωγείς παιχνιδιών για τα παιδιά μας. είναι ενάμιση χρόνο σήμερα από όταν είχαμε καινούρια οδηγία ωστόσο πάλι σήμερα είμαστε εδώ όπως και πέρυσι όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο πρόεδρος να μιλάμε για το ίδιο θέμα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και φέτος τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. γιατί; γιατί έχουμε κρίση και όταν έχουμε κρίση οι γονείς θέλουν να αγοράσουν παιχνίδια δεν έχουν χρήματα θα πάνε στο τμήμα εκείνο της αγοράς που έχει παιχνίδια κατώτερης ποιότητας. όταν όμως έχουμε παιχνίδια κατώτερης ποιότητας έχουμε τρία προβλήματα πρώτον το τμήμα εκείνο της αγοράς δεν έχει γνώση των κανόνων δεύτερον δεν έχει προσωπικό τρίτον δεν υπάρχουν οι έλεγχοι. άρα εξακολουθούμε να είμαστε απροστάτευτοι και όπως όλοι ξέρουμε και όλοι δεχόμαστε τα παιδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε και όπως εσείς κύριε επίτροπε πολύ σωστά είπατε είναι οι περισσότερο ευάλωτοι πολίτες. λοιπόν σας παρακαλώ απαντήστε για το ce που είναι η εγγύηση ασφάλειας σας παρακαλώ κύριε επίτροπε δώστε απαντήσεις στην πράξη ώστε του χρόνου ούτε εσείς να είστε εκεί ούτε εμεί να είμαστε εδώ να κάνουμε την ίδια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Στήλερ, δύο λεπτά. Το θέμα της ασφάλειας των παιχνιδιών είναι πολύ σημαντικό για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παιχνιδιών και οι γονείς πρέπει να, έχουν, να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι ε, τα παιχνίδια που αγοράζουν για τα παιδιά τους είναι απόλυτα ασφαλή. Εδώ βρισκόμαστε στις 11.30 να μιλάμε για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να το καταλάβω. Τι πρέπει επιτέλους να γίνει. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή ποιες εταιρείε παιχνιδιών που διανέμουν οι πουλάνε παιχνίδια ε, ε, διώχθηκαν διότι είχαν χρησιμοποιήσει παράνομα το ΣΥ σε ό,τι αφορά την επιτήρηση της αγοράς. Τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη δεν, δεν επαρκούν, δεν είναι καθόλου επαρκή σε τοπικό επίπεδο λόγω περικοπών προϋπολογισμού και για άλλους λόγους ε, ε, ε, υπονομεύεται και δεν εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Τι παρακολούθηση γίνεται ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη προστατεύουν τα παιδιά από τη χρήση επικίνδυνων παιχνιδιών και τι γίνεται με το θέμα της επιτήρησης και της εποπτείας της αγοράς. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία πρέπει να αποσύρονται άμεσα από την αγορά. Υπάρχει ε, ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επιθεωρητών της αγοράς στα διάφορα κράτη-μέλη Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα επικίνδυνα προϊόντα θα αποσύρονται από την αγορά μόλις διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα. Ελπίζω ότι το 2011 επιτέλους θα κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο απόλυτα ασφαλή προϊόντα. Ο κ. Ζεγκέντη είναι ο μόνος ε, αγωγητής μέσω της δικασίας Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα παιδιά είναι το μέλλον μας, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουν ασφάλεια στην ε, πρώιμη παιδική του ηλικία. Οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς δεν είναι παρά μόνο ένα τμήμα ε, αυτές τις διαδικασίες. Είναι σημαντικό να ξεπίσουμε τους ε, κανόνες. Είναι σημαντικό να διενεργούνται σωστοί έλεγχοι και σε περιπτώσεις παραβίασης να θεσπιστούν κάποιες κυρώσεις. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για θεγινά παιχνίδια. Εγώ είμαι πατέρας και πολύ συχνά έχω την αίσθηση ότι τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά μου ε, είναι πολύ κακής ποιότητας και πολλούνται πραγματικά μαζικά. Θα πρέπει να απαγορευθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλη. Για ένα λεπτό. Α, ο κύριος Κέλλη. Ε, ε, ε, μίλησα για το θέμα αυτό πέρσι και όπως και οι άλλοι ομιλητές ε, ε, βρίσκομαι εδώ για να διαπιστώσω ότι πέρασε άλλος ένας ε, χρόνος και πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να διαπιστώνουμε ότι ζημιώνεται η υγεία των παιδιών ή πεθαίνουν παιδιά λόγω αυτών των επικίνδυνων παιχνιδιών. Ε, τα ποστά των καρκίνων αυξάνονται ιδιαίτερα μεταξύ μικρών παιδιών και πολλοί έχουν την εντύπωση ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της έκθεσης σε τοξικές ε, ουσίες, για παράδειγμα ε, σε πολυκυκλικούς υδρογονάφρακες. Επίσης, γι' αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τοξικές αυτές ουσίες σε ένα στο ελάχιστο ε, κατόφλι. Ε, θα πρέπει να το πράξουμε επιτέλους και να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιχνίδια που συμβούν τα παιδιά μας είναι ασφαλή για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, να απαντήσω στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν και να υπενθυμίσω εκ νέου ότι η οδηγία θα εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις από τον Ιούλιο του 2011. Οι υποχρεώσεις για τις χημικές ουσίες θα εφαρμόζονται από τον Ιούλιο του 2013. Είπα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου ότι για την Επιτροπή η εφαρμογή των νέων κανόνων από πλευράς όλων των εμπλεκομένων πλευρών αποτελεί προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο μια αυστηρή νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αυτή δεν θα είναι αποτελεσματική ποτέ αν δεν εφαρμόζεται σωστά. Γι' αυτό είμαι πεπισμένο ότι τα κράτη-μέλη διαδραματίζουν και μπορεί να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα προϊόν που έχετε στο Ρότερνταμ, στην ε, Κωνσταντσα, στο αύριο θα είναι στην Πολωνία ή στη Λισαβόνα χωρίς άλλο έλεγχο. Άρα αυτό που δίνει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές είναι η εμπιστοσύνη στην καλή λειτουργία της εποπτείας της αγοράς. Στο γεγονός δηλαδή ότι αν κάποιος προσπαθήσει να περάσει επισφαλή προϊόντα θα υποστεί κυρώσεις και τα προϊόντα που είναι επικίνδυνα θα αποσυρθούν από την αγορά. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και τις επιχειρήσεις. Εκείνες που τηρούν τους κανόνες και πληρώνουν το κόστος θέλουν να ξέρουν ότι δεν υφίσταται τον αθέμητο ανταγωνισμό αυτό που παράγουν επικίνδυνα προϊόντα με μικρότερο κόστος μη τηρώντα τους κανόνες. Συνθετικά, η πρόκληση για τους, την ασφάλεια των καταναλωτών είναι level playing field, ισότιμη μεταχείριση και καλή εποπτεία. Γι' αυτό η Επιτροπή το 2011 θα εξετάσει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα πολιετών τους χαρακτήρα για την εποπτεία της αγοράς που θα επιτρέπει τον εντοπισμό των δράσεων που πρέπει να, έχουν, να υλοποιηθούν στην, σε μακρά περίοδο και να έχει τα κατάλληλου τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για να υπάρξει ένα ε, καλό επίπεδο ε, ε, αυστηρών ελέγχων σε συνέπεια με τις παρεμβάσεις των κρατών μελών. Επιπλέον θέλω να αναγγείλω ότι η πρόθεσή μου είναι να οργανώσω μια εκδήλωση του 2011 ίσως ταυτόχρονα με τη θέση ισχύ της στο Ρότερνταμ μαζί με τις Ολλανδικές Αρχές για να δούμε ε, πώς θα οργανωθεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης ε, για την υλοποίηση των νέων ε, επιταγών της οδηγίας. Ό,τι αφορά το σήμα Ευρω... ECE e, που ήταν στο κέντρο της ακρόασής μου στο Κοινοβούλιο πριν την, ε, λάβω την εμπιστοσύνη και που ήταν ένα θέμα συζήτησης και σε άλλες ακροάσεις που είχα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Θέλω να επιθυμίσω ότι το σήμα CE δεν πιστοποιεί την ποιότητα, αλλά μόνο την τήρηση κάποιων κανόνων. Ένα πιστοποιητικό είναι πιστοποιητικό τήρηση κανόνων, όχι πιστοποιητικό ποιότητα. Ένα σήμα ποιότητα μπορούμε να το σκεφτούμε μόνο για το μέλλον, όπω είπα πολλέ φορέ. Ήδη είναι πολύ μεγάλη δουλειά η υλοποίηση του σήματος E και να υποφύγουμε την καταχρηστική χρήση του όπως πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει με προϊόντα που προέρχονται και εκτός Ευρωπαϊκή, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά προωθώντας και αυξάνοντας και βελτιώνοντας το σήμα. Εγώ δεν είμαι αντίθετο ε, με το να εξετάσουμε στο μέλλον και την υιοθέτηση ενός σήματος ποιότητας, όχι όμως τώρα, είναι πρόημο. Προβλέπεται άλλωστε στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων. Τώρα, για, το, για τη βυσφενόλη που περιλαμβάνεται στα μπιμπερό των παιδιών δεν είναι παιχνίδι, δεν καλύπτεται, το μπιμπερό δηλαδή είναι παιχνίδι, δεν καλύπτεται από την οδηγία, αλλά ήδη έχει αποσυρθεί από την αγορά του συγκεκριμένου προϊόν. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και ευχαριστώ τους κύριους και τις κύριες βουλευτές που έφεσαν τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας και πάλι αύριο το πρωί στις 8.30. Καλό σας βράδυ.